Καλησπέρα σας συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να σας καλωσορίσω όλους στην συνεδρίαση της Επιτροπής TAX 3 μετά τις ακροάσεις για τη διάσταση των τρίτων χωρών στην καταπολέμηση των φορολογικών ε, ποινικών αδικημάτων της φοροαποφυγής και φοραπάτης την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της, οργανώνοντας ακρόαση για τις σχέσεις με την Ελβετία σε φορολογικά ζητήματα. Θα έχουμε ένα και μόνο πάνελ, με μια σειρά από παρουσιάσεις από τους εμπειρογνώμονές μας, τους προσκεκλημένους μας, που θα επικεντρωθούν στη γενική προσέγγιση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Θα δούμε επίσης τη νομική θέση και κατάσταση των ε, όσων καταγγέλουν, των καταγγελόντων, τις σχέσεις τους που μπορεί να έχουν ε, με, τις τραπεζικές, με τα τραπεζικά ιδρύματα και τι σχέση μπορούν να έχουν τα ιδρύματα αυτά με, τη λεύκανση, με, την, με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Όσο για τους ομιλητές του πάνελ είναι ο κύριος Γκίτερ Κίσελ, καλώς ήρθατε, ο οποίος είναι τμήματάρχης των επιζήμιων ε, φορολογικών πρακτικών, της υπηρεσίας επιζήμιων φορολογικών πρακτικών ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Ταξούτ, ο κύριος Έλμερ, Κάπου εδώ είναι μάλλον. Καλώ ήρθατε κύριε Ρούντολφ Έλμερ. Είστε καταγγέλων από την ε, Ελβετία. Κύριε Έλμερ, δουλέψατε σε τράπεζα στο, στη Julius Bar από το 1980 μέχρι την απόλυσή σας, την απομάκρυνσή σας από το 2002. Αποκαλύψατε απόρριτα τραπεζικά έγγραφα στο Wikileaks με λεπτομερείς ε, περιγραφές του τι έκανε η Γιούλιου στις νήσους Κέιμαν. Τον ε, Ιανουάριο του 2011 καταδικαστήκατε στην Ελβετία για την παραβίαση του νόμου περί απορρίτου, τραπεζικού απορρίτου. Ε, η υπόθεσή σας θα συζητηθεί σε δημόσια ακρόαση από το Μοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας στις 10 Οκτωβρίου. Η δημόσια ακρόαση πρόκειται να είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, διότι αφορά το θέμα του κατά πόσον το ελβετικό τραπεζικό απόρριτο μπορεί να ισχύει και εξωεδαφικά ή όχι. Και μετά να καλωσορίσω τον κύριο Ανδρέας Φρανκ, πρώην τραπεζικό και ειδικό για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος από τη Γερμανία, θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι η ΕΕΔ ε, προσεκλήθη σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για να παρουσιάσει το πώς έχουν εξελιχθεί οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας για τη διμερή συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς όμως δεν βρίσκονται σήμερα εδώ επειδή ούτως ή άλλως θεωρούν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ λεπτή, λεπτό σημείο. Οι δύο επικεφαλείς διαπραγματευτές ε, δεν ήρθαν λοιπόν, αλλά δεν μας εμποδίζει αυτό να συζητήσουμε όσα εμείς θεωρούμε σκόπιμα. Ίσως γραπτός να τους ενημερώσουμε κατόπιν για το ποιες είναι οι δικές μας ανησυχίες πώς θα εργαστούμε τώρα. Κάθε ομιλητής θα έχει το πολύ 7 λεπτά για την παρουσίασή του. Μετά τις παρουσιάσεις θα έχουμε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Κίφελ να μας παρουσιάσει την δική του εισήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσω τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας σε φορολογικά θέματα. Στην άμεση φορολογία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερες σχέσεις σε δύο τομείς με την Ελβετία. Το ένα είναι η διοικητική συνεργασία και ο άλλος τομέας είναι η επιζήμια, ο επιζήμιος φορολογικός ε, ανταγωνισμός. Ε, εγώ θα μιλήσω μόνο για τη διοικητική συνεργασία, γιατί το άλλο ε, είναι στα χέρια άλλων. Στο πρωτόκολλο στις 27, είναι από τις 27 Μαΐου 2015 και αφορά ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και Ελβετίας, μεταξύ φορολογικών αρχών. Το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 από το, από το 5 ε, χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία δέουσας επιμέλειας ε, για τη συλλογή φορολογικών πληροφοριών ε, επιλογαριασμών που τηρούνται άμεσα ή έμεσα από Ελβετούς υπηκόους και υπηκόους της Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες αυτομάτως ανταλλάσσονται μεταξύ της χώρας συλλογής και της χώρας κατοικίας του πραγματικού ιδιοκτήτη. Ε, η πρώτη τέτοια ανταλλαγή έγινε το Σεπτέμβριο του 2018, ε, τους τελευταίους μήνες. Η συμφωνία συνάδει με το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή ε, πληροφοριών και λογαριασμούς σύμφωνα με τον ΩΣΑ και τους G20, την πρότυπα, κοινά πρότυπα αναφορών. Επίσης προβλέπεται η παροχή ε, πληροφοριών μετά από αίτημα ε, για την καλύτερη λειτουργία των φορολογικών αρχών στην Ελβετία και στα κράτη-μέλη. Και έτσι περνώ στην ομάδα ε, του κώδικα δεοντολογίας. Ε, δεν είναι δεσμευτικό όργανο. Πρόκειται για τον εντοπισμό επιζήμιο, επιζήμιου ανταγωνισμού στα φορολογικά θέματα. Ε, υπάρχει, αφορά τα κράτη-μέλη. Αλλά η, αρχή αυτή ε, μπορεί να επεκταθεί σε συναφή εδάφη και γειτονικέ χώρες. Το 2010 ο κώδικας διοντολογίας αποφάσισε να ανοίξει διάλογο με τις γειτονικές χώρες Λίχτενστάιν και Ελβετία ε, με βάση τις αρχές του κώδικα. Μετά από 7 χρόνια διαλόγου, τα κράτη-μέλη και η Ελβετία ε, έκαναν κοινή δήλωση τον Οκτώβριο του 2014. Σύμφωνα με την κοινή αυτή δήλωση, η Ελβετία πρέπει να καταργήσει πέντε επιζήμια φορολογικά καθεστώτα και να απέχει από την εισαγωγή νέων ε, μέτρων αντικατάστασής τους. Από τη μία πλευρά, αφού η Ελβετία θα συμμορφωθεί ε, προς το κοινή δήλωση, τα κράτη-μέλη δεν θα εφαρμόζουν αμυντικά μέτρα και αμυντικές πρακτικές σε σχέση με αυτά τα καθεστώτα. Η ε, πραγματοποίηση των, ε, του περιεχομένου της κοινή δήλωσης θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού και θα μειώσει τον επιζήμιο ανταγωνισμό. Το Ιούνιο του 2016 το Ελβετικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε μεταρρύθμιση του νόμου που θα καταργούσε τα πέντε επιζήμια καθεστώτα. Όμως σε ένα δημοψήφισμα που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου του 2017 οι Ελβετοί απέρριψαν τη φορολογική μεταρρύθμιση. Έτσι λοιπόν όλο το νομοσχέδιο ε, που συμπεριλάμβανε και την κατάργηση θα έπρεπε να αντικατασταθεί με, ναι, από νέα πρόταση. Σε διμερές επίπεδο, μετά το δημοψήφισμα, οι ελβετικές αρχές ανέλαβαν να συμπεριλάβουν την κατάργηση των πέντε καθεστώτων στη νέα τους νομοθεσία. Μία επιστολή εστάλει στον πρόεδρο της ομάδας δεοντολογίας και επιβεβαίωσε τη δέσμευση. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ είχε αποφασίσει το 2016 η ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιου... κατήρτιζε έναν κατάλογο μη συνεργαζομένων ε... ε φορολογικών ε, αρχών ε, και η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μια εξέταση και αξιολόγηση των 92 φορολογικών συστημάτων που επελέγησαν η Ελβετία συγκαταλεγόταν σε αυτά τα φορολογικά συστήματα, τα επιζήμια που τα μη συνεργαζόμενα και συμπεριελήφθη στο εγχείρημα. Επειδή η Ελβετία ήδη είχε ε, πει ότι θα καταργούσε τα πέντε μέτρα, η Ελβετία δεν εκλήθη να αναλάβει δέσμευση για δεύτερη φορά. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ λοιπόν έβαλε την Ελβετία μεταξύ των τρίτων χωρών και των φορολογικών του συστημάτων που έκαναν τις σωστές δεσμεύσεις στο λεγόμενο παράρτημα 2. Και αυτές οι χώρες δεν θα ήταν στον κατάλογο των μη συνεργαζομένων φορολογικών συστημάτων με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκρίνονταν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Το 2017 η ελβετική κυβέρνηση παρουσίασε νέα πρόταση στο Κοινοβούλιο που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η προηγούμενη σε σχέση με την κατάργηση των πέντε επιζημίων ε, καθεστώτων. Φαίνεται ότι το Ελβετικό Κοινοβούλιο ψήφισε την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή στις 28 Σεπτέμβρη, το νέο νόμο. Σήμερα τα πράγματα έχουν ως εξή. Η Κομισιόν είναι σε στενή επαφή με την Ελβετική Διοίκηση. Αναμένουμε να ενημερωθούμε πλήρως έφθετο χρόνο για τη νέα νομοθεσία και να πάρουμε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για να την εξετάσουμε. Να εξετάσουμε το νομοσχέδιο κομισιόν, θα ενημερώσει την ομάδα δεοντολογίας με τις απατούμενες πληροφορίες, ώστε η ομάδα να ε, πάρει μια απόφαση βάσει στοιχείων σχετικά με το αν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις η Ελβετία, για να μην συμπεριληφθεί ως φορολογική διοίκηση που δεν συνεργάζεται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Keeping to the time limit, although... Θα σας ζητήσω να κρατάτε το χρονικό όριο, παρότι έχουμε ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα. Κύριε Έλμαρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση θα κάνω κάποιες ε, δηλώσεις για τις οποίες δεν είμαι περήφανος, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Here we go. Now I would like to touch on these points I mentioned uh, in the introduction. Θα σας ε, παρουσιάσω τα σημεία αυτά της εισαγωγής. Πρώτα απ' όλα, η καταγγελία ενός εγκλήματος αποτελεί έγκλημα στην ε, Σουηδία, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ελβετία. Στην Ελβετία, συγγνώμη. Στην ε, Ελβετία. Ε, αυτό σημαίνει κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό θάνατο για τον κατακέλλοντα. Ε, γνωρίζω πολλές περιπτώσεις και πρόσφατα οι καταγγέλτες ε, κατηγορούνται και καταδικάζονται για διάφορους λόγους. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι ένα σημαντικός κλάδο, σημαντική κλάδη στην Ελβετία Αυτή που βλέπετε εδώ ε, στη, με κόκκινο χρώμα έχουμε το Swiss Payment Center, το ελβετικό κέντρο πληρωμών στο περνό της Ρήχης. Ε, πραγματοποιεί πληρωμές εντός της Ελβετίας. ώστε να αποφεύγει την υποβολή πληροφοριών που απαιτεί το σύστημα SWIFT διότι το SWIFT είναι το σύστημα των ΗΠΑ. Υπάρχει ένα ε, σύστημα πληρωμών στην Ελβετία, στο Ιζήριχη. Το δεύτερο που επισημαίνω είναι ότι παλιότερα ε, ε, μπάνκερ του ελβετικού στρατού χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μη οικονομικών περισσότερων στοιχείων. Ανθεί λοιπόν ο κλάδος αυτός στην Ελβετία και νοικιάζουν διάφορους χώρους, ε, διάφοροι, διάφορα άτομα σε μπάνκερ όπως αυτά. Πώς προστατεύει αυτούς τους βασικούς κλάδους και τους εκπροσώπους τους η Σουηδία. Να σας υπενθυμίσω τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει κατά βάση είναι ότι ουσιαστικά οι έρευνες απορρίπτονται. Οι αιτήσει για έρευνες. Ε, για παράδειγμα, είχαμε έρευνες κατά τις UPS ε, ε, του κ. Όσπολ απορρίφθηκε. Ορισμένες έρευνες δεν ξεκινούν καν. Η Ελβετία πραγματοποιεί βρώμικες συμφωνίες ώστε να κλείνουν οι έρευνες αναφέρομαι στην υπόθεση HSBC στη Γενέβη. Το θυμάστε όπου το κατάστημα της Γενέβης βρισκόταν υπό έρευνα λόγω μη ε, ε συμμετοχής ε, σε θέματα ε, φοροδιαφυγής και ξεπλήματο μαύρου χρήματος. Έγινε μία λοιπόν συμφωνία για προς τιμού 40 εκατομμυρίων. Ε, δηλαδή ουσιαστικά απαλλάσσεται κανείς από μια υπόθεση ε, νομοποίησης ε, εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με κάποιο πρόστιμο. Υπάρχει μια ελαφρία τιμωρία για οποιονδήποτε κατηγορούμενο για οποιοδήποτε, οποιοδήποτε αδίκημα στον τομέα. Με μια ελαφρία τιμωρία. Υπάρχει ένα παράδειγμα ενό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στη Γενέβη, ο οποίο καταδικάστηκε ε, ε, ως βοηθός στη δημιουργία εταιριών offshore για την κάλυψη της προέλευσης ε, ε, κονδυλίων και λογαριασμών και έλαβε ουσιαστικά μία καταδίκη με αναστολή, τρίμηνη και πλήρωσε τα δικαστικά έξοδα. Η προστασία των καταγγελτών στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, παρότι έχουν προσπαθήσει να τη δημιουργήσουν από το 2003 ε, συναντά ε, διαρκείς ε, καθυστερήσεις. Εξακολουθεί να μην υπάρχει. Το επόμενο είναι τα αντίπεινα κατά καταγγελτών, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ακραία. Καταγγέλτε στην Ελβετία ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό θάνατο στην Ελβετία. Να σας δώσω και κάποιες ε, εικόνες ε, για το απόρριτο στην υπόθεση ε, για, για την υπόθεση Έλμερ εναντί Swiss Bank Secrecy. Το 2005 αποφασίστηκε στη Ζηρίχη ότι τα όσα κατασχέθηκαν στο δικό μου σπίτι στην Ελβετία δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο έρευνα από τι ελβετικέ αρχέ, από τι ελβετικέ φορολογικέ αρχέ. Η αιτία που έδωσαν ήταν ότι είναι ασυνήθιστο να βρει κανεί δεδομένα με μια κατοικών έρευνα για μια τράπεζα στα νήσου Κέιμαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα οι φορολογικέ αρχέ. Εγώ υπέβαλα διάφορε καταγγελίε ε, για Ελβετού πελάτε στην Ελβετία, διότι είμαι ακτιβιστή. Όλε αυτέ όμω οι καταγγελίε απορρίφθηκαν με την ε, αιτιολογία ότι εγώ δεν έχω υποστεί προσωπικά κάποια ζημιά δεν δόθηκε καμία σημασία στα στοιχεία αυτά ούτε από τις ελβετικές αρχές ούτε από τις διοπτικές αρχές. Ε, ε χρησιμοποιήθηκαν όμως από άλλες χώρες όπως η ΕΠΑ, η Γερμανία και ούτω καθεξής. Το, γραφείο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο της Εισαγγελίας, στο οποίο απευθύνθηκα το 2009 μετά από την υπόθεση Wikileaks, η Guardian, στον Ηνωμένο Βασιλείο, δημοσίευσε ένα άρθρο με ονόματα Μεξικανών εμπορών ναρκωτικών και λοιπόν το γραφείο λοιπόν, το Ομοσπονδιακό Γραφείο της εισαγγελία, ε, στο οποίο εγώ έδωσα στοιχεία, απάντησε μετά από 10 ημέρες και είπε ότι δεν έχουν καμία σχέση αυτά με την Ελβετία. Έλαβα μία απάντηση τεσσάρων γραμμών ουσιαστικά. Η τράπεζα είχε λάβει μία επιστολή πέντε σελίδων που τους εξηγούσε ε, οπότε, εντάξει, δεν υπήρχε καμία σχέση με την Ελβετία. Στο Ομοσπονδιακό ε, Δικαστήριο της Ελβετίας ε, εγώ έλαβα καταγγελίες από το Συμβούλιο είπα ψέματα για τη δική μου υπόθεση η εποπτική αρχή των χρηματοοικονομικών αγορών, μια ανεξάρτητη αρχή, πραγματοποιεί έρευνες, αλλά μου είπαν ότι δεν θέλουν να τις δημοσιοποιήσουν στη δική μου περίπτωση. Η ουσία είναι λοιπόν είναι ότι στην έρευνα κατά της ε, Γιούλες Μπέρ, ε, τους εκπροσώπους της και ε, την έδρα του στην Ελβετία έχει ακυρωθεί. Συγγνώμη, ο πρόεδρος, πρέπει να επιταχύνουμε. Έχετε ξεπεράσει ήδη τα 8 λεπτά. Στην επόμενη διαφανή ήθελα να σας αναφέρω ε, ποιες είναι οι, δικαστικές, οι νομικές αιτίες που οδηγούν ε, σε offshore. Ουσιαστικά η εισαγγελία ε, ρωτά ε, ε, τον κατηγορούμενο αν έχει ας πούμε, ένα τράστιο στο Denver του λέει ότι αυτό δεν θα ερευνηθεί. Είχαμε και οργανωτικούς λόγους με τις ε, τηλεπικοινωνίες ε, στην περίπτωση της, των Βερμούδων ε, ανακατεύθυναν κλήσεις ώστε να φαίνεται σαν να υπάρχει δραστηριότητα στη, στη Βερμούδα, στις Βερμούδες. Τώρα έχουμε τις ελβετικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Μιλήσαμε για τα καθεστώτα, τα οποία πρέπει να καταργηθούν, αλλά υπάρχουν νέα ελβετικά αντίμετρα, κατά την άποψή μου. Έχουμε το Patent Box, ε, ε, κίνητρα έρευνα και ανάπτυξη στα καντόνια, την μείωση των φορολογικών συντελεστών ε, σε κεφάλαια, διάφορα προνόμια και τη μείωση των, της φορολογίας στα καντόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Το βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια που πως πραγματοποιήθηκε από... Βλέπετε ότι οι φόροι για τις εταιρείε μειώνονται. Η Γενέβη έχει 24% σήμερα και τώρα κατεβαίνει στο 13%. Η Γενέβη είναι ένα χρηματοοικονομικό κέντρο και κέντρο καταναλωτικών προϊόντων. προϊόντων. Η Βασιλεία επίσης ε, ουσιαστικά οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται σε επίπεδο τέτοιο που εξακολουθεί να είναι δυνατή η προσέλκυση και η διατήρηση των επιχειρήσεων εκείνων που θέλει ουσιαστικά να φορολογούνται δικαίως όσα. Ε, αφήνουμε αυτή τη διαφάνεια γιατί μιλάμε για, τους, ε, για τα δύο μέρη. Ε, εδώ σας παρουσιάζω την κατάσταση στη δική μου οικογένεια. Έχω υποστεί απειλές και εκβιασμό, ψυχολογική βία Ε, έχω στραφεί επανειλημμένως κατά της εφημερίδας που ε, έγραψε κατεμού. μου. Ε, βρέθηκα σε κράτηση υπό περιορισμό για αρκετές μέρες. Η κόρη μου έκανε απόπειρα αυτοκτονίας διότι της απαγγέλθηκαν κατηγορίες ο αδελφός μου γιατί έχουμε ακόμα την ευθύνη των συγγενών. Ο αδελφός μου εργάζεται για την αστυνομία και δεν μπορούσα πλέον να μιλήσω μαζί του διότι του ανέφεραν ότι διακινδυνεύει η θέση του διότι είναι αδερφό μου και ούτω καθεξής. Συνεχίζεται λοιπόν η κατάσταση αυτή, το κυνήγι μαγισσών που γνωρίζουμε κατά των καταγγελτών στην Ελβετία. Τι λέω λοιπόν εδώ, ότι εξακολουθώ να είμαι ακτιβιστή και εξακολουθώ να μάχομαι. Δεν υποχωρώ και ελπίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου θα εμφανιστώ στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και θα, ε, θα απαιτήσω να ε, Πραγματοποιήσουμε μια δήλωση για το απόρριτο των ελβετικών τραπεζών. Δεν είναι θέμα δικό μου προσωπικό πλέον, αφορά το θέμα του απορρίτου των ελβετικών τραπεζών. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο κύριος Φρανκ. Όπως σας εξηγήσαμε, δεν είμαι Ελβετός, είμαι Γερμανός και από τη Νέα Υόρκη δούλεψα μετά στην Ελβετία και καταλαβαίνετε ότι η μέθοδος εργασίας μου είναι να είμαι πολύ πρακτικός και ρεαλιστής και έτσι θα κάνω και την παρουσίασή μου. Μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις διμερείς συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετία. Η στρατηγική των Ελβετών δεν το θέλουν αυτό πριν το Brexit, τον Μάρτιο του 2019 διότι θέλουν να συνεχίσουν διαλέγουν ό,τι τους βολεύει. Τα επιζήμια φορολογικά συστήματα λοιπόν, αυτό που εδώ και χρόνια επικρίνει ο ΣΑ. Και σε αυτές τις δημοτεύσεις καταλήξαμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Οι Ελβετοί έκαναν δημοψήφισμα, ε, θα κάνουν μάλλον δημοψήφισμα να ρωτήσουν τους πολίτες και θα πάρει χρόνο για να λάβουν τη σωστή απόφαση οι Ελβετοί. Στην Ελβετία ε, θέλουν να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Έχουν και μια έκφραση γι' αυτό στα, στα γερμανικά της Ελβετίας. Και αυτό κάνουν και με τις συμφωνίες τους. Ε, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Θυμάμαι όταν ε, ξεκίνησε η συμφωνία δίωξης της UBS, η Ελβετία, η ελβετική κυβέρνηση, ακολούθησε την ε, λεγόμενη πολιτική του λευκού χρήματος ε, και μετά τα ε, εφάρμοσε στον ελβετικό χρηματοοικονομικό τομέα. Και το ελβετικό τραπεζικό απόρριτο υπάρχει ακόμα. Είναι πολύ εύκολο να κρύψει κανείς το πραγματικό ιδιοκτήτη σε μια άλλη δικαιοδοσία. Και μετά από Αμερικανό πολίτη μπορείτε να μετατρέψετε κάποιο σε πολίτη της Μπαχάμας και στέλνουν τις πληροφορίες εκεί, άμα θέλουν και γελάνε κιόλα. Ε, πάνε όλα στον κάλαθο των αχρήστων και δεν γίνεται και τίποτα. Αδύνατο να ερευνηθεί. Βάσει του δικτύου μας για τη φορολογική δικαιοσύνη, η Ελβετία είναι η χειρότερη χώρα ως προς το χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό απόρριτο. Και παρόλα αυτά είναι ε, το μεγαλύτερο κέντρο ε, υπεράκτειας, θα λέγαμε, ε, δυνατότητας να κρύβει κανείς χρήμα. Η Ελβετία παραμένει το στο μοντέλο όλων των ε, φορολογικών παραδείσων με, με συστήματα φορολογικού απορρίτου και τραπεζικού απορρίτου. Όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν. Εάν δείτε την τελευταία φετινή έκθεση του Ωσάλε, την ε, όλη ιστορία με λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να δούμε τις επιμέρους πληροφορίες. Υπάρχει σχετική έκθεση, μπορείτε να τη διαβάσετε. Η Ελβετία ε, θα πρέπει να δεχτεί περισσότερο τι καταγγελίε των καταγγελότων και να καταπολεμήσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και θα πρέπει όσοι λειτουργούν παρα, παρανομίε στην Ελβετία να πληρώσουν πρόστιμα. Από δικηγόροι μέχρι τραπεζίτε που δεν ε, έχουν καμία ποινική δίωξη προ στιγμή. Μόλι είπε ο γειτονά μου ότι ε, έχει διωχθεί ποινικά. Και ο φάκελό του είναι γνωστό στον Όσα. Είναι ε, μια έκθεση που έχει γίνει και έχει καταρτιστεί πλήρω και δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να αλλάξει κανείς και να κλέψει και σε αυτό το σύστημα, αλλάζοντα την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη. Στο άλλο γράφημα λέει ότι όταν δεν σας αρέσει το μήνυμα σκοτώνετε τον αγγελιοφόρο. Αυτό εξηγεί. Δηλαδή πώς οι επιζήμιες πρακτικές απορρίτου στην ε, Ελβετία που από το πολιτικό σκέλος από την ε, Βουλή και τα κόμματα. Το 2016 στη Σουηδία ψηφίστηκε αλλαγή, ψηφίστηκε αλλαγή στο νόμο για τις υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών, ώστε να ε, προστατεύουν τους καταγγέλλοντες και ε, από το εξωτερικό και να δέχονται τα αποδεικτικά τους στοιχεία. Στη Γερμανία, υπεύθυνο γι' αυτό, ας πούμε, είναι το Υπουργείο Οικονομικών όμως στην Ελβετία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι νόμοι χρησιμοποιούνται για να πάψουν να ομιλούν όλοι αυτοί που έχουν κάτι να πούν εντός της χώρας και εκτός. Και μάλιστα τη δράση την αναλαμβάνει ο, από τους διάδικους ο εισαγγελέα. Ο, ενάγ, ο εναγόμενος, όχι ο ενάγων. Ε, επιβάλλεται ε, να υπάρχει ένα μητρό πραγματικής ιδιοκτησίας. Διότι, ας πούμε, λόγω, χάρη στο δικό μα γερμανικό νόμο για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, η πραγματική ιδιοκτησία μιας εταιρεία εφόσον τύχει να είναι στην Ελβετία, μπορεί να οδηγήσει στη Ζηρίχη για να πρέπει να μιλήσει κανεί με του ομολόγου του εκεί, αλλά τελικά να μην παίρνει καμία απάντηση. Κάτι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μου κυβέρνηση κάτι θέλει να κάνει για να προστατεύσει και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όλου αυτού του ανθρώπου που θέλουν να δώσουν πληροφορίε για το Μητρό των Πραγματικών Ιδιοκτητών τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόζουν αποφάσεις του Ελβατικού Δικαστηρίου. Αν πάρει κανείς πρόστιμο στην Ελβετία, υποχρεώται να το πληρώσει. Ισχύει και στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να πάυσει. Ε, πρέπει να ακολουθήσουμε το αμερικανικό μοντέλο, το νόμο του Ομπάμα που έλεγε ότι δεν αναγνωρίζονται η σχετική νόμη ευθύνη ε, της Ε, Το λέμε αυτό άγρα δικαιοδοσίας, ε, την ε, άγρα της σωστής δικαιοδοσία για να μην έχει κάνει ευθύνη. Από τη Βρετανία μπορεί κανείς να πάει στην Ελβετία και να είναι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει. Κάτι ακόμα που βρίσκω πολύ σημαντικό είναι το αν θέλει κανείς να θολώσει τα νερά ε, και να προλάβει την εποπτεία. Ε, μπορεί με τις αρμόδιες αρχές στην Ελβετία, αυτές που ασχολούνται με το ξέλιμα του βρώμικου χρήματος, να κάνει αυτό που τον βολεύει, γιατί μιλάμε για αυτορυθμιζόμενους φορείς. Πληρώνουν για αυτούς ιδιώτες και μου συνέβη και εμένα αυτό. Προστατεύουν τα μέλη τους ε, με κάθε τίμημα. Και ακόμη και οι μυστικές πληροφορίες, οι απόρριτες πληροφορίες που δίνονται στις επόπτες είναι γνωστές τα μέλη και μπορεί να οδηγήσουν και σε μηνύσεις για ε, δυσφήμιση ε, κατά αυτού που δίνει τις πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, είναι σχεδόν ανύπαρκτη η εποπτεία, έστω πολύ αδύναμη. Και ε, ακόμη και εταιρείε ε, κρυπτονομισμάτων στο καντόνι του Τσούχ, ας πούμε, ε, καμαρώνουν ότι είναι στο κέντρο της παγκόσμιας παραγωγής και στην Ομοσπονδιακή μας Βουλή και από τις Ηνωμένε Πολιτείες ομολογός μας κοίταξε τις αποκεντρωμένες εταιρείες και των στον κόσμο και είδε ότι είναι η πιο τα πιο ισχυρά κέντρα στην Ελβετία, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκεί ο νόμο. Ε, και δεν χρειάζεται και τραπεζικό λογαριασμό. Όλα αυτά λοιπόν μα διαφεύγουν. Δεν είναι περίεργο που η Ελβετία το χρησιμοποιεί αυτό το όπλο, αυτή τη νέα τεχνολογία, για να καλύψει παράτυπο χρήμα και με άλλους τρόπους. Για να συνοψίσω, ε, νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχει προοπτική για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, θα πρέπει οι υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργοί να περάσουν την Ελβετία σε έναν μαύρο κατάλογο, σε αρνητικό κατάλογο για την έλλειψη συνεργασίας της. Και στις επισκέψεις μου, το επιβεβαίωσε και όσα, η Ελβετία θα πρέπει να είναι στον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών με στρατηγικά ε, κενά και ελλείψεις για την καταπολέμηση του ξεπλήματος δρόμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να κάνει, γιατί και σε 20 και σε 30 χρόνια, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Φρανκ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη βέβαια θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε 30 λεπτά περίπου, όχι παραπάνω. Λοιπόν, τέσσερα λεπτά, ένα λεπτό δηλαδή η ερώτηση, τρεις η απάντηση. Αρχίζουμε με τους συνεισηγητές. Ο κυρίος Νίντερμαέρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πέτερ, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους. Εγώ ε, εστιάζω στην Κομισιόν Ήμουν μέρος της αποστολής πάνω στην Ελβετία. Ξέρω την κατάσταση λοιπόν και τα πορίσματά μας, αλλά και τα αποτελέσματα της ειδική ομάδας για τα χρηματοοικονομικά. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ποινές ε, δεν είναι αποτρεπτικές προκειμένου περί ξεπλήματος, ε, δεν οδηγούν στην αλλαγή και οι συναλλαγές είναι μικρές ε, που αναφέρονται, είναι λίγες. Υπάρχει πρόβλημα με την δέουσα επιμέλεια και δεν παρακολουθούνται οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ερωτώ την Κομισιόν, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα ή είμαστε σε στασιμότητα. Και να αναδιατυπώσω αυτό που είπε ο κύριος Φράνκ. Ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελβετίας στον κατάλογο των χωρών που κάνουν ξέπλυμα. Δεύτερον, μετά την αποστολή μας στη ΣΥΠΑ ακούσαμε ότι οι Αμερικανικές αρχές είναι πολύ ικανοποιημένε με το τραπεζικό πρόγραμμα της Ελβετίας. Φαίνεται ότι πιστεύουν ότι οι ελβετικές τράπεζες κάνουν πολύ καλή δουλειά για τις αμερικανικές φορολογικές ε, αρχές για να αντιμετωπίζουν τους φορολογουμένους τους οι Αμερικανοί. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ελβετικών τραπεζών και ευρωπαϊκών αρχών για σε σύγκριση με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ ελβετικών τραπεζών με τις αμερικανικές αρχές. Ε, ο κύριος Κίσελ να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίτερ Μάιερ για την ερώτηση. Φοβάμαι ότι μερικώς θα απαντήσω στην ερώτησή σας μόνο, γιατί εγώ ε, μιλώ για τις, τα φορολογικά θέματα, για την ταξούτ. Δεν μπορώ να μιλήσω για το ξέπλυμα χρήματος και τη συνεργασία εκεί που ρωτήσατε. Τώρα, για την ανταλλαγή πληροφοριών είπα ε, τα σχετικά. Το αναθεωρημένο πρωτόκολλο έχει ολοκληρωθεί, το 2014 τέθηκε σε ισχύ και η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα. Άρα λοιπόν το σύστημα λειτουργεί, αλλά δεν μπορώ να σας πω εδώ και τώρα πόσο καλή είναι η ποιότητα και αν αξίζει τον κόπο και αν είναι επαρκείς οι πληροφορίες, γιατί πρέπει να αναλύσουμε ε, την ουσία των πληροφοριών που μας ε, δίνονται, αλλά δεν είχαμε χρόνο για να το κάνουμε αυτό μέχρι τώρα, οπότε δεν μπορώ και να δώσω μια ουσιαστική απάντηση που να αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και το ποιόν της. Ε, μιλήσατε και για το γκρίζο κατάλογο. και εδώ. Ε, ναι, μεν είμαι αρμόδιο σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση για τον απλό λόγο ότι ο νόμος που μεταρρυθμίζει τα, τις φορολογίες ε, μόλις την περασμένη εβδομάδα πέρασε. Εμείς ε, δεν αξιολογούμε τα νομοσχέδια στην ομάδα δεοντολογίας, άρα πρέπει να περιμένουμε να μας ενημερώσουν οι ελβετικές αρχές για τον νόμο πλέον που έχει ψηφιστεί. Γιατί δεν εξετάζομαι τα νομοσχέδια πριν περάσουν από το Κοινοβούλιο. Για δύο λόγους. Ε, η φορολογική διοίκηση του κράτους ε, θα λάβει κυρίαρχη απόφαση, οπότε δεν μπορεί να παρεμβαίνει η δικιά μας ομάδα δεοντολογίας σε αυτή τη διαδικασία και δεύτερον θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι πολλές φορές ε, γίνονται τροπολογίες ε, στα νομοσχέδια για λόγους ε, πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οπότε δεν έχει νόημα. Για αυτούς τους δύο λόγους η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας εξετάζει και αξιολογεί μόνο ψηφισμένα νομοσχέδια, νόμους πλέον. Οπότε και εν προκειμένου πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε την τελική ενημέρωση από τους ε, Ελβετούς συναδέλφους. Μάλιστα. Ο κύριος Κόφορτ, συνεισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα προς την Επιτροπή για την ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσετε. Αυτά που δεν έχετε πάρει ακόμα από τους Ελβετούς. Μπορείτε να, δεν μπορείτε να σχολιάσετε, αλλά μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε για τη συμφωνία με την Ελβετία και ήμουν υπεύθυνο ηγετή για το θέμα αυτό από το Κοινοβούλιο. Είμαι πολύ περίεργο. Ε, μπορείτε να αξιολογήσετε κατά πόσον παρακάμπτουν τι υποχρεώσει του για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών φορολογικών πληροφοριών. μπορούν να το κάνουν αυτό απευθεία οι τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διότι έχει σημασία για το τι κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν ε, σημαντικό να δούμε το πνεύμα τη συνεργασία μα ξανά και για την προστασία των καταγγελόντων. Ε, Υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο πρέπει να προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη συμφωνία με την Ελβετία κάποια ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ανθρώπων αυτών στον ιδιωτικό τομέα επίση, όταν αφορά την ασυλία του, την νομική του αρρωγή και άλλα πράγματα. Κατά την άποψή σα, πρέπει να υπάρξουν ενδεχομένω διεθνή πρότυπα για την προστασία των ανθρώπων αυτών. Πρόσφατα στη Δανία με την Danske Bank είχαμε ένα θέμα καταγγελίας ε, με έναν ε, πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που έκανε κάποιες καταγγελίες και τώρα φοβάται για την σωματική του ακαιρεότητα, για την οικογένειά του, γιατί έκανε κάποιες καταγγελίες. Η ανωνυμία του μάλιστα εκτέθηκε από την ίδια την τράπεζα στα, στη δημόσιο, ε, σε δημόσιο, στη δημόσια γνώση και δημοσιεύτηκε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πώς μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερη προστασία των καταγγελόντων. Ο κύριος Έλμερ. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρωτάτε. Νομίζω είναι εύκολη η δουλειά. Απλή μάλλον. Πρόσφατα είχα πάει στην ε, Σερβία και άκουσα για το σχετικό νόμο προστασίας των καταγγελόντων εκεί. Κατά την άποψή μου, είναι ε, σημαντικό γιατί έχουν εκπαιδεύσει τους εισαγγελείς, τους δικαστές που ασχολούνται με τις υποθέσεις καταγγελιών βάσει του νόμου αυτού και έχουν αρκετές επιτυχίες από τις 30 υποθέσεις που παρουσιάζονται 27 από τη δεύτερη και τρίτη μέρα εκδίκαση έχουν δικαστική απόφαση. Ε, δικαστική απόφαση και για την προστασία μάλιστα του καταγγέλλοντος. Ο νόμος υπάρχει λοιπόν. Θα σας έλεγα να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το νόμο. Αντιγράψτε τον. Ο Στίβεν Κόεν από τις Ηνωμένε Πολιτείε έχει μελετήσει και εκείνο αυτόν τον νόμο προστασίας των καταγγελόντων. Είναι πραγματικά ένα από τα υψηλότερα δίχτυα προστασία που παρέχονται. Ευχαριστούμε πολύ. Επιτροπή. Ω προ την ερώτησή μου, μου είπατε ότι θα αξιολογήσετε την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνετε από την Ελβετία. Και επίση, ήθελα να σα ρωτήσω εάν μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρακάμπτουν τι υποχρεώσει του για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμε για φορολογικού σκοπού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό ακούσαμε ότι κάνουν ε, με τη δημιουργία νέων ε, συστημάτων. Έχετε λοιπόν κάποιο είδου άποψη που θα μπορούσατε να τη μοιραστείτε με το Κοινοβούλιο. Ναι, το κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι ήταν σχόλιο αυτό που είπατε. Θα φροντίσω να μεταβιβάσω το μήνυμα αυτό. Τεχνικώς σας ενδιαφέρει τι είδους ε, πληροφορίες έχουμε μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, δηλαδή τράπεζε των κρατών μελών ε, που επικοινωνούν μεταξύ του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τι παίρνει αυτέ τι πληροφορίε, δεν έχει τι λεπτομέρειε. Τα βλέπουμε όταν ε, συναντιόμαστε και συνεδριάζουμε με τα κάτι μελη όταν έχουμε μαζί του ανταλλαγή πληροφοριών και τότε αξιολογούμε τη γενική ποιότητα πληροφοριών. Θα φροντίσω να το μεταβιβάσω και όταν έχουμε την απαραίτητη αξιολόγηση θα σα ενημερώσω. Ω προ την ποιότητα λοιπόν και το κατά πόσον ε, υπάρχουν ε, τάσεις να παρακάμπτονται υποχρεώσεις. Κύριε Έλμερ, ναι, μία δήλωση ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. εγώ έχω δουλέψει 8 δικαιοδοσίε και μου αρέσει η πρακτική προσέγγιση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δουλεύει μόνο εάν ο πελάτη έχει ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του. Τότε γνωρίζει τι γίνεται και ποια είναι η ταυτότητά του. Αν όμω έχουμε μια εταιρεία σε κάποιο ε, άγνωστο μέρος ε, και οι διευθυντές οι διευθυντές, οι γραμματείς, οι δικηγόροι ε, και όλοι αυτοί είναι πρόσωπα πίσω από τα οποία δεν υπάρχει καμία πραγματική ταυτότητα ε, από την άποψη αυτή, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα βήμα, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να ψάχνουμε ψήλο στάχυρα, έναν άγνωστο στο δρόμο. Έχουν ε, κάνει έτσι τα συστήματά τους οι εταιρείε αυτές, περάκτιες, ε, ε συστήματα για να κρύβουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Και έτσι κρύβονται. Ναι. Ναι, έχω δει και πραγματικά έγγραφα όπου Ελβετική Τράπεζα ξέπλυνε βρώμικο χρήμα αλλάζοντας ταυτότητα συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή, εάν Αμερικανός πολίτης στείλει λεφτά στο Χονγκ Κόνγκ μέσω τριών εταιριών, επανέρχεται χωρίς να υπάρχει παραμικρή ε, σχέση με τον πραγματικό ιδιοκτήτη και να μπορεί να βρεθεί. Ε, άλλοι πληρώνουν 30% παραπάνω και αυτός κάνει ό,τι έκανε συνήθως. Οι τράπεζες τα γνωρίζουν αυτά. Γίνεται εκ προθέσεως και είναι μεγάλη, ε, μεγάλη πηγή κέρδους. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια εδώ πέρα, τότε αξίζει τον κόπο. Η Ομοσπονδιακή Βουλή τον Απρίλιο του 2017 τροποποίησε τον γερμανικό νόμο για, την, ε, για το ξέπνιμα βρώμικου χρήματος με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που άρχισε να εφαρμόζεται. Είναι πολύ δύσκολο οι φορείς να καταγράψουν στοιχεία όταν τα ονόματα λιώνονται και κρύβονται. Διότι ξαφνικά το σύστημα κρύβει τα ονόματα που γίνονται ανώνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά. Πρέπει να ρίξουμε και μια δεύτερη ματιά, είναι βέβαιο. Για να δούμε πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητες και στην ε, φοροδιαφυγή. Μου κάνει έκπληξη, με συγκλονίζει που ακούω όλα αυτά που ακούω, το πώς η Ελβετία παρακάπτει τους κανόνες που υπάρχουν και τις διατάξεις της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε πρέπει να ρίξουμε μια ματιά σε μεγαλύτερο βάθος. Τώρα, για τις ερωτήσεις. Εμείς ήμασταν σε, πρόσφατα σε μια αποστολή στη Λετωνία, η οποία αυτό έγινε στο πλαίσιο του σκανδάλου ABLV στη Λετωνία όπως είναι γνωστό, τεράστιες ε, ποσότητες χρημάτων ε, έχουν μεταφερθεί από μη ε, κατοικούς, μη διαμένοντες και τελικά σε άλλους προορισμούς. Η Λετωνία δεν ήταν ο τελευταίος, ο τελικός προορισμός. Και μεταξύ αυτών των δικαιοδοσιών που έλαβαν τα χρήματα αυτά, που ήταν ο προορισμό αυτών των χρημάτων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η Ελβετία. Μιλάμε για χρήματα που ήρθαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλε χώρε μέσω του λετονικού τραπεζικού συστήματος χάρη στη χαλαρή επιτήρηση εστάλησαν έτσι μεταξύ άλλων στην Ελβετία. Θέλω να μάθω το δικό σας σχόλιο. Αληθεύει ή όχι, έχετε κάποια εκτίμηση του μεγέθους αυτών των ε, κονδυλίων, αυτών των χρημάτων, το δεύτερο. Μελετάμε αυτή τη στιγμή ένα νομοθετικό πακέτο της φορολόγησης των ψηφιακών εταιριών ένα νομοθέτημα αποτελεί μια πρόταση επιβολή σε βραχή πρόθεσμων φορολογικών μέτρων, ώστε να γίνει κάτι με αυτέ τι ψηφιακέ εταιρείε πριν όσα τελικά καταλήξει μια κοινή θέση, κάτι απίθανο. Θέλω να μου πείτε την άποψή σα. Πώ πιστεύετε ότι θα αντιδράσει η ελβετική κυβέρνηση σε όλα αυτά, Τι ρόλο πιστεύετε ότι παίζει στο, στο αρμόδιο φόρουμ του ΩΣΑ υποστηρίζει μια τέτοια ιδέα ή αντιτίθεται σε αυτήν. Ευχαριστούμε. Για την πρώτη ερώτηση, ποιος θα θέλει να απαντήσει. Okay, so Mr. Elmer, about the... Κύριε Έλμαρ, για το μέγεθος, ε, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκτός μικροφώνου μίλητης. Υπάρχουν ενδείξεις. Αλλά ο τομέας, ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας στην Ελβετία έχει μεγάλες τράπεζες και ανθεί. Γι' αυτό ανθεί, επειδή υπάρχει τεράστια εισρωή χρημάτων, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αλλά οι ενδείξεις είναι υπαρκτές. Ότι η Ελβετία τα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον τραπεζικό του τομέα. Οι τεράστιες τράπεζες, αυτές αναφέρομαι, όχι στις μικρές. Κατά την απόψή σα, τι θέση θα κρατήσει η Ελβετία όσον αφορά τη φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών. Επιτροπή. Δεν είμαι εμπειρογνώμων, αλλά αυτό μπορώ να σας πω από τις προσωπικές μου γνώσεις είναι ότι η Ελβετία στις συζητήσεις του ΩΣΑ διατηρεί μια επιφυλακτική, προσεκτική στάση. Αναλύει τα πάντα πολύ προσεκτικά, λεπτομερώς Συγγνώμη, ρωτάω ο μιλητή. Αυτά γνωρίζω, λέει ο μιλητή. Ωραία, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Όπω εξήγησα, οι αρμόδιες αυτέ αρχέ τη Ελβετία δεν λειτουργούν. Δεν έχουν φτιαχτεί για να λειτουργούν. Γι' αυτό το λόγο, όταν εμεί συνομιλούμε με αρμόδιες αρχέ, οι πληροφορίε που μας δίνουν ε, είναι αναξιόπιστες. θα έπρεπε να έχει κανεί άμεση πρόσβαση, όχι να μιλά μέσω άλλων οι οποίοι φιλτράρουν τις πληροφορίες. Ίσως θα έπρεπε να πω κάτι στην Κομισιόν. Έχουμε αυτές τις υποθέσεις με τις τράπεζες, την Danske Bank, την ING και τις άλλες τράπεζες. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Στην τις ε, τρίτες χώρες και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα ε, χειριζόμαστε όπως θα έπρεπε ε, βάσει των όσων λέει η Task Force. Είμαστε μέλος της Task Force για τη χρηματοδοτική δράση. Αξιολογούμε την Κομισιόν, ενώ θα πρέπει να αξιολογούμε τα κράτη-μέλη και καταλήγουμε σε πρότυπα τελικά μόνο. Ευχαριστώ. Εφτά ε, ε, ευρωβουλευτές είναι γερμανόφωνοι και ε, δύο από τους μιλητές μας. Να σας ρωτήσω λοιπόν, Έλμερ και Φρανκ, μετά από αυτά που μας είπατε, και ιδιαίτερα ο κύριος Φρανκ είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο τέλος. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση το σύστημα δεν λειτουργεί και είναι σχεδιασμένο για να μην λειτουργεί. Από την πολιετή σας πείρα, τι θα συμβουλεύατε στην Ευρω... την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ε, κινήσεις πρέπει να κάνει ε, για να ασκήσει πιέσεις και να λειτουργούν τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι αρχές. Και μια ερώτηση στον κύριο Κίσελ από την Κομισιόν. Κύριε Κίσελ, δεν κατάλαβα γιατί δείχνετε τόση κατανόηση στην Ελβετία. Είπατε θα ε, εξετάσετε το νόμο, θα δείτε τι ε, θα γίνει, τι πληροφορίες ε, δίνουν, τι δεσμεύσεις θα αναλάβουν. Η ΕΠΑ έδωσε μέχρι τέλος του 2018 μια σκληρή προθεσμία για να συμμορφωθούν Παρθένη, Νήσι και όλοι οι άλλοι Κάιμαν. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο με την Ελβετία. Τους πιάνουμε με το γάντι εδώ και χρόνια. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να περιμένετε το νόμο και να δείτε αν μας εξυπηρετεί. Γιατί να μην δείτε το status quo και να πείτε στο τέλος του χρόνου θα μπει στον κατάλογο. Και αν η Ελβετία φέρνει ένα νόμο που δικαιολογεί την απόσυρση από το, την απάλληψη από τον κατάλογο να απαλληφθεί. Γιατί δεν κάνετε έτσι. Ο κύριος Φρανκ και ο κύριος ε, Κίσελ. Άσκηση πίεση στην Ελβετία. Αυτό θα έπρεπε να το κάνει η ειδική ομάδα ε, για τα χρηματοοικονομικά. Ε, θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις, ε, τις πληροφορίες που έχουν. Το, το φόρουμ είναι το, ο σωστός, ε, είναι η ενδεδειγμένη ομάδα για να παρουσιάσει αυτές τις ε, πληροφορίες. Επίσης, υπάρχουν δυνατότητες που πρέπει να είναι γνωστές στον κόσμο. Ε, ε, χρειάζεται αξιολόγηση της Ελβετίας ε, που θα καταλήγει στη διαπίστωση ότι δεν συνεργάζεται. Και έτσι θα μπουν στον γκρίζο ή στο μαύρο κατάλογο. Ένα βασικό θέμα είναι οι φορολογικές συντελεστές, οι χαμηλοί. Πριν από πέντε μέρες ε, στη Ζηρίχη έγινε γνωστό ότι εταιρείε στη Ζηρίχη ε, πληρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια λιγότερους φόρους λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών και των αντίμετρων που έχουν προβλέψει και εφαρμόζουν. Για τα αντίμετρα, εδώ το θέμα είναι να δούμε με έρευνα και ανάπτυξη. Ποιε είναι οι δαπάνε για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα. Τι επιτρέπεται να πάει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει, υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Οι, οι ε, μεγάλες εταιρείες ε, ε, έχουν δυνατότητα να κινηθούν ευέλικτα. Εμείς Πρέπει να ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσα κεφάλαια θα διοχετεύονται στην έρευνα για την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η Ελβετία πρέπει να βρει τη θέση στο μαύρο κατάλογο. Ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Οι Αμερικανοί, γιατί έγινε συζήτηση για τους Αμερικανούς και πώς αντιμετωπίζουν τους Ελβετούς, ε, υπάρχουν Αμερικανοί, υπάρχει και ένας εμπειρογνώμων ο οποίος ε, έχει την εποπτεία των τραπεζών και είναι σε καλύτερη θέση με το σύστημα που έχουν. Πάντως και η Ευρώπη μπορεί να κάνει το ίδιο, παρόλο που δεν ε, έχουμε τον ε, έλεγχο του δολαρίου, αυτό είναι στα χέρια των Αμερικανών, θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή λογαριασμό σε δολάρια για να γίνονται πληρωμές σε δολάρια στις ΗΠΑ ασκούν ε, πιέσεις στις τράπεζες και λένε ότι δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές, ε, μπορεί να το πει, σε δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πει ότι αν δεν ε, συμμορφώνεται η Ελβετία θα επιβληθούν κυρώσεις παρόμοιες. Είναι κρίμα που τα λέω αυτά για τους Ελβετούς, αλλά λέω την αλήθεια, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και είναι και πολλοί στην Ελβετία που συμμερίζονται τις απόψεις μου και δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση σήμερα στην, στην Ελβετία. Ε, Κομισιόν, μπορώ να απαντήσω και εγώ στα γερμανικά, αφού ο κύριος Ευρωβουλευτής ερώτησε στα γερμανικά. Μπορώ. Εντάξει. Κύριε Βουλευτά, είπατε γιατί δείχνουμε τόση κατανόηση και ε, ε, εμείς ποιοι είμαστε εμείς. Ε, καταρχήν πρέπει να δούμε τις αρμοδιότητες. Επίσης, η επιζή, ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ο κώδικας δεοντολογίας και τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία ε, ασκούν πιέσεις μεταξύ ομολόγων και υπάρχουν οι πιέσεις για να ε, βελτιωθούν τα φορολογικά συστήματα όταν είναι επιζήμια και η Κομισιόν έχει ένα τεχνικό ρόλο. Εμείς ε, βοηθούμε, επικουρούμε. Τώρα, γιατί πάνε τόσο αργά τα πράγματα. Ναι, αλλά γιατί δεν τους βάζετε στον κατάλογο, αφού κάνατε πρόταση για κατάλογο. Ναι, να εξηγήσω γιατί κινούμεθα αργά. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελβετία δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί. Ο κατάλογος, ε, τι κατάλογος είναι, είναι κατάλογος των φορολογικών διοικήσεων που δεν συνεργάζονται. Φορολογικές διοικήσεις ε, που δεν συνεργάζονται. Μπορεί να ήταν λάθος ε, έτσι όπως ονομάσαμε τον κατάλογο, αλλά οι φορολογικές διοικήσεις που δηλώνουν πρόθυμες να κάνουν αλλαγές και να πάνε ε, στη σωστή πλευρά δεν πάνε στο μαύρο κατάλογο. Και το 2014 ήδη η Ελβετία δήλωσε ότι είναι πρόθυμη. Δεν θέλω ε, να υπερασπιστώ την Ελβετία, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αλλά το 2016 πρέπει να πούμε ότι η Ελβετία ε, έδωσε τα παραδοτέα της για πρώτη φορά και ο νόμος ε, δεν πέρασε λόγω του δημοψηφίσματος το 2017 όχι γιατί ήταν άδικα τα μέτρα, αλλά γιατί ο κόσμος δεν ήταν ε, σύμφωνος ε, με τα μέτρα ε, που αφορούσαν του νόμου για τη χρηματοδότηση. Μετά την αποτυχία, μετά την αποτυχία της πρώτης προσπάθειας, μετά το δημοψήφισμα, η Ελβετία πάλι είπε ότι ήταν πρόθυμη να τηρήσει τα υπεσχημένα και υπέβαλε νέα νομοθετική πρόταση ε, κινούνται λίγο αργά, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Ελβετία. Αλλά καταρχήν συνεργάζεται με βραδύτητα, αλλά συνεργάζεται η Ελβετία. Γι' αυτό. Δεν ακούστηκε η παρέμβαση. Ε, αυτό θα το αποφασίσει η ομάδα δεοντολογίας στο τέλος του χρόνου. Η, η Ελβετία όμως ε, δεν είχε νόμο. Ναι, αλλά το 2014 η Ελβετία ήταν πρόθυμη να αλλάξει τα πράγματα. Οι εθελοντικά δηλαδή δεσμεύτηκαν πριν υπάρξει ο κατάλογος. Ε, νομίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ε, η, κυρία Λαπεκορέλα που είναι η πρόεδρος της ομάδας διοντολογίας ε, το ξέρει αυτό. Ε, μπορείτε να τη ρωτήσετε. Η απόφαση επίσης δεν θα ληφθεί από την Κομισιόν, η σχετική απόφαση, αλλά από την ομάδα του κώδικα δεοντολογίας. Ε, και εκείνοι θα το κρίνουν αυτό το ζήτημα. Η δε απόφασή τους θα ληφθεί τον Ιανουάριο του χρόνου. Μπορείτε να ρωτήσετε αυτό το πράγμα ε, στην κυρία Πεκορέλα. Καταλαβαίνω την ενόχλησή σας. Ευχαριστώ. Βολφ Κλίντς. Συνεχίζω και εγώ στα γερμανικά. Πριν από 30 χρόνια, για πολλά χρόνια εργαζόμουν στην Ελβετία και ε, τότε δεν μου έκρυβαν οι Ελβετοί ότι ε, αξιοποιούν το τραπεζικό απόρριτο για πολλά και διάφορα κόλπα και συμφωνίες και με άλλους Ελβετούς και με ε, τρίτους. Και επίσης ε, προσήλκησαν και Γερμανούς να μεταφέρουν τα χρήματά τους ε, στην Ελβετία με ευνοϊκά καθεστώτα. Εν τω μεταξύ άλλαξαν κάποια πράγματα και εγώ εξεπλάγει ακούγοντα όλα αυτά από τους τρεις ειδικού γιατί νόμιζα ότι εδώ και καιρό τα πράγματα είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι τέλεια. Ε, αυτή η αλλαγή είναι και πολιτισμική ε, η πολιτισμική αλλαγή δεν γίνεται μια ανοιχτή. Και αναρωτιέμαι, τι θα κάνουμε. Σχέσεις ε, με την Ελβετία σε φορολογικά θέματα και στη μάχη κατά του ξεπλήματος χρήματος. Αυτό είναι ο τίτλος. Δηλαδή έχουμε φορολογικά θέματα αφενός και ξέπλυμα χρήματος. Στα φορολογικά θέματα, εκεί το θέμα εν πωλήση ε, είναι Ε, η φορολογική παράδειση και ή ο αθέμητος φορολογικός ανταγωνισμός. Δεν ξέρω αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και εμείς τόσο καθαροί. Γιατί αν δω το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα νησιά της Μάνχης, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γιβραλτάρ και λοιπά και λοιπά ε, και, και εμείς έχουμε μεγάλες διαφορές. Η Ελβετία ως αποκεντρωμένο σύστημα ε, μπορούν να έχουν φορολογική αυτονομία των καντονίων. Ε, αλλά έχουν ενίο σύστημα προσδιορισμού. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια βάση προσδιορισμού του φόρου εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και δεν θα τα καταφέρουμε και ποτέ έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Οπότε, δεν νομίζω ότι είμαστε οι αναμάρτητοι για να ρίψουμε το, τον λίθο. Τώρα για το ξέπλυμα του χρήματος. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Μιλάμε για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με το τραπεζικό τομέα και το χρηματοοικονομικό τομέα. Αλλά το ξέπλυμα χρήματος έχει και άλλα. Τα, την τέχνη, τα ναρκωτικά, τα κίνητα. Και αν σκεφτώ και τη δικιά μου τη χώρα, τη Γερμανία, μιλάμε για τριψήφια νούμερα σε δισεκατομμύρια τα οποία μ, ξεπλένονται μέσω αυτών των καναλιών και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να προσδιορίσουμε ε, ποσοτικά το πρόβλημα, να το δημοσιοποιήσουμε και να το καταπολεμήσουμε. με την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, ότι δεν μπορεί να γλιτώσει έτσι εύκολα η Ελβετία, αλλά πώς. Νομίζω ότι η Ελβετία γενικά σε επίπεδο οικονομίας εξαρτάται πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίκλειστη χώρα όπως ακούσαμε και δεν μπορεί χωρίς ε, να έχει σωστέ οικονομικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναπτυχθεί και εκείνη καλά. Άρα λοιπόν τις διμερείς συμφωνίες που έχουμε θα τις χρησιμοποιήσω όμω. μοχλό και θα πούμε αν μέχρι τότε και μέχρι τότε δεν βελτιωθούν τα πράγματα τότε ε, οι προτιμησιακές συμφωνίες θα τεθούν εκτός ισχύως. Γιατί όλα αυτά, ότι θα μπει στον κατάλογο, θα βγεις από τον κατάλογο, δεν είναι τόσο πιστικά. Όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε με, το, με τις τράπεζες, ε, μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε ανάλογους μοχλούς πίεσης. υπάρχουν πολλές, πάνω από 100 διμερείς συμφωνίες και η ερώτηση είναι, αυτές οι διμερείς συμφωνίες ε, αποτελούν μοχλό πίεσης. Να πούμε δηλαδή ότι αν δεν συνεργαστείτε, τότε θα ανασταλεί θα ανασταλούν αυτές οι συμφωνίες. Η άσκηση πίεση είναι ένα θέμα, αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται και καθοδήγηση, ένα προσανατολισμό. Τι προσανατολισμό θα τους δώσουμε. Μπορεί κανείς να πει ότι ε, τα κέρδη των επιχειρήσεων θα πρέπει να φορολογούνται με συντελεστή 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι είναι κάτω, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 15. Δεν έχει σημασία τώρα το νούμερο. Αυτό που είναι όμως κάτω από αυτό αποτελεί επιζήμια φόρο αποφυγή. Όχι, δεν είναι ανόηση αυτό, διότι έτσι δίνεται ένα προσανατολισμό και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολύ απλή μέθοδο για να δείξετε τι περιμένετε από, εκείνους. Κάτω από το αν πέσει ο συντελεστής, τότε αναλαμβάνεται δράση. Δεν θα καταφέρετε ποτέ να, το να εφαρμοστεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένουν τα κράτη-μέλη στην εθνική τους κυριαρχία σε φορολογικά θέματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο ορατό μέλλον να εισαχθεί κοινό ίσως φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις και στα 27 κράτη-μέλη. Αποκλείεται. Πρέπει να το δεχτούμε. Η Apple τιμωρήθηκε γιατί δεν πλήρωνε αρκετούς φόρους στην Ιρλανδία. Τι έκανε η Apple. Πήγε στο Jersey όπου πληρώνει λιγότερο από 1%. Ορίστε, βρήκε τη λύση. Εμεί υποκρινόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε τη λύση, αλλά εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε το ίδιο κακοί με την Ελβετία. Δεν έχουμε προοδεύσει καθόλου. Πρόεδρο, ε, ευχαριστώ, David Coburn. Θέλατε να πείτε κάτι. Σφάιν, συγγνώμη. Μην παραπονεθείτε όμως ότι σας αφήνουμε να μιλήσετε, Σβέν. Ε, και εγώ στα γερμανικά θα μιλήσω, αφού πολλοί μιλούν γερμανικά εδώ και θα τα καταλάβετε και καλύτερα. Απευθύνομαι κυρίως στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Εδώ από το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα επιζήμιου ανταγωνισμού. Παλιό το θέμα. Το Ελβετικό Κοινοβούλιο με το νομοσχέδιό του προέβησε διορθώσεις. Και θέλω να μου πείτε, στη διαδικασία αυτή του νομοσχεδίου πώς συμμετείχατε. Σας ρώτησε αν οι Ελβετοί σας ρώτησαν αν οι νέες ρυθμίσεις ε, είναι συμβατές με τις ε, προϋποθέσεις της Ένωσης. Το ρωτώ αυτό γιατί αφενός τα ελβετικά καντόνια ε, ήδη είναι ε, τα πιο ευνοϊκά εις ό,τι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Και τώρα στη, στην κατάταξη θα έχουν ακόμα πιο ευνοϊκή θέση. Επίσης, όταν ε, κάποια αέδρα πάει στην Ελβετία, ε, ε, ε, αντιμετωπίζεται προνομιακά. Έχουμε ειδικό φορολογικό και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις ευρεσιτεχνίες. Ε, υπάρχει έκπτωση ε, στη φορολογία κερδών. υπάρχει επίσης η αρχή της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης μιας θηγατρικής, μιας παραφιάδας μιας εταιρείας. Ε, θα ήθελα να μου πείτε, αυτά τα μέτρα όλα τα έχετε αναλύσει. Μπορείτε να τα αναλύσετε και πώς θα ε, περιορίσετε αυτόν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντωμεταξύ έχει πάρει και άλλα μέτρα. Έχουμε ένα μητρό που είναι κοινό ε, ε, μεταξύ των 28 για, τους, ε, για όσους δραστηριοποιούνται ε, οικονομικά. Μπορεί, υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελβετία. Η Ελβετία δεν έχει μηχανισμούς ε, για φορολογικές για φορολογική στήριξη. Εμείς έχουμε, εσείς ως Κομισιόν τους πιέσατε ώστε να λάβουν παρόμοια μέτρα. Επίσης, στην ανταλλαγή πληροφοριών ομαδικές ερωτήσεις και αιτήματα μπορούν να γίνουν μόνο ε, βάσει της ε, διπλής φορολόγησης, ενώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Συμφωνίας για τη διπλή φορολόγηση, που δεν καλύπτει το παρελθόν. Οπότε, πολλοί που έκαναν φοροδιαφυγή στη Γερμανία Αξιοποιώντα το φορολογικό καθεστώ της Ελβετίας, δεν μπορούν πια να εντοπιστούν. Ε, επίσης, ε, υπάρχουν θέματα που δεν εμπίπτουν στην ε, ομάδα δεοντολογίας, αλλά είναι ενωσιακό δίκαιο. Ε, υπάρχουν ε, φορολογικές αποφάσεις που μπορούν να δοθούν στην Ελβετία ούτω ώστε να συμμορφωθούν προς τις αποφάσεις. Επίσης, ε, υπάρχουν ε, ε, πολλές φορές διαδικασίες ασυμβίβαστες με την αρχή της ελεύθερης διακίνησης. Εκεί δεν θα πρέπει να γίνει ευθυγράμμιση. Ε, ε, ε, επίσης, στο φόρο κύκλου εργασιών υπάρχουν διαφορετικές προθεσμίες υποβολής των στοιχείων και έτσι γίνονται διακρίσεις υπέρ των μεγάλων εταιριών. Και μια ερώτηση για την Κομισιόν. Έχετε αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχετε ώστε στα πλαίσια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων ε, σε διμερές επίπεδο και ε, στα πλαίσια των άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ε, είχατε, αξιοποιήσατε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις ελλείψεις και τι μέτρα λάβατε ούτως ώστε οι ελλείψεις αυτές να καταργηθούν. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσει η Κομισιόν γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά. Ευχαρίστω, ε, λέει ο μιλητή, να τα απαντήσω γραπτό. Μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία ή θα τα στείλετε γραπτό ενδεχομένω καλύτερα. Μπορώ να δώσω μια σύντομη προφορική απάντηση. Αν θέλετε να δώσω και γραπτή. Εγώ θα ακολουθήσω την πρόταση του Προέδρου. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τις διμερείς συμφωνίες, ήδη είπα στην αρχή ότι εγώ είμαι υπεύθυνο για τη ε, Γενική Διεύθυνση Τάξου για τα φορολογικά θέματα και όχι της ε, υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτό είναι θέμα διοργανικό και νομίζω ότι δεν θα ε, μπορούσα εγώ να σας απαντήσω εδώ. Ε, πρέπει, όπως είπε ο Πρόεδρος, να απευθυνθείτε στην, εξωτερική, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις ε, διμερείς συμφωνίες για ενημέρωση. Τώρα, για τις ε, πιο λεπτομερείς ερωτήσεις. Αν μας ρώτησαν για το νομοσχέδιο το 2017 όχι, δεν μας ρώτησαν εμάς για το νομοσχέδιο αυτό οι Ελβετοί, διότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις εμπίπτουν στην ε, εθνική αρμοδιότητα και στην εθνική κυριαρχία του κάθε κράτους, το οποίο διαμορφώνει το φορολογικό του δίκαιο όπως ξέρει καλύτερα. Αυτόνομα δηλαδή έδρασαν οι Ελβετοί. Από την άλλη μεριά ρωτήσατε τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα την αναλύσω, βέβαια θα αναλύσω με τα μέτρα που προβλέπει πρέπει να ελέγξουμε και να δούμε αν τα πέντε επιζήμια καθεστώτα που έπρεπε να καταργηθούν όντως καταργήθηκαν, αυτό είναι σχετικά εύκολο να γίνει. Παράλληλα όμως θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε αν συνεχίζεται η διαδικασία εισάγοντας νέα επιζήμια καθεστώτα. Γιατί η Ελβετία στην κοινή δήλωση ε, ανέλαβε τη δέσμευση να καταργήσει τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα χωρίς να τα αντικαταστήσει με άλλα επιζήμια ε, για τα patent box, τα φορολογικά ευνοϊκά καθεστώτα για τις ε, και τις εκπτώσεις. Εδώ υπάρχουν διεθνή πρότυπα και εκεί θα στηριχθούμε για να κρίνουμε το νέο νόμο των Ελβετών. Είπατε επίσης για ε, το 150% έκπτωση για έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό ε, προβλέπει, ε, αυτό γίνεται για τις ε, επενδύσεις και την προσέλκυση κεφαλαίων στην έρευνα και ανάπτυξη. Εμείς αυτό το θέλουμε. Και επίσης υπάρχει και ειδική έκπτωση για την έρευνα και την ανάπτυξη και στον, στην κοινή βάση προσδιορισμού του φόρου. Ε, αν τους πιέσαμε να ε, υιοθετήσουν ένα ευρωπαϊκό μητρό. Ε, εδώ μιλώ... Εδώ, επαναλαμβάνω, έχουμε τη, τη διεύθυνση για τα φορολογικά θέματα και είμαστε περιορισμένοι στα επιζήμια καθεστώτα. Δεν κάνουμε εναρμόνιση, ελέγχουμε τα αλλά η ομάδα αυτή ε, της δεοντολογίας εξετάζει αν εισάγονται φορολογικά καθεστώτα που δημιουργούν διακρίσεις και προνόμια. Ε, τώρα, αν θα έπρεπε να υπάρχει ένα, δημόσιο μητρό, αυτό δεν είναι θέμα της, της ομάδας δεοντολογίας. Ε, Ε, για την ε, ενημέρωση, δεν πιέσαμε, η, η Ελβετία είναι μέλος του ΟΣΑ και στους κόλπους του ΟΣΑ είναι και μέλος ε, της ομάδας εργασίας για φορολογικά επιζήμια μέτρα. Ε, υπάρχει εκεί πρόβλεψη ανταλλαγής δικαστικών αποφάσεων, παράλληλη δέσμευση όπως ε, ε, υπάρχει και για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ενωσιακό επίπεδο. Και επειδή προβλέπεται αυτό, η Ελβετία στα πλαίσια του ΩΣΑ πρέπει να κοινοποιεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων ε, στις χώρες του ΩΣΑ. Προβλέπεται ανταλλαγή πληροφοριών για τα rulings, για τις αποφάσεις αυτές επιφορολογικών θεμάτων. Ε, εδώ και καιρό υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης για το πώς προχωρούμε. Δεν ξέρω τώρα που έχουν προχωρήσει. Πριν από καιρό ήμουν υπεύθυνο γι' αυτό και είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες. Με έκπληξη άκουσα ότι δεν, προχώρησαν, ε, δεν προχώρησε η συνεργασία όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις του κυρίου Βουλευτή. Αν ε, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις θα μας τις θέσετε και θα απαντήσουμε με γραπτή διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ήδη, κράτησε περισσότερο η συνεδρίασή μας. Οι διερμηνείς θα μας εγκαταλείψουν στις 10. Έχουμε ελάχιστα λεπτά, David Coburn. Πριν φύγουν όλοι, σε ό,τι αφορά τους καταγγέλλοντες. Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να ρισκάρουν και στα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να έχουμε επιπόλους ε, καταγγέλλοντε από ό,τι θέλουν και ό,τι του κατέβει να πηγαίνουν, να παίρνουν ένα φωτοτυπικό και να διαδίδουν πράγματα και να σφυρίζουν στη σφυρίχτρα του, όπω λέμε από τα αγγλικά και την αγγλική λέξη. Βλέπουμε ότι εδώ πολύ λίγοι ξέρουν από επιχειρήσεις οι καταγγέλλοντε να πάνε στα δικαστήρια και σε κάποιε περιπτώσει να περιφθεί και η υπόθεσή του. Εγώ πήγα και στην Επιτροπή Paradise Papers και παρά την τεράστια κατακραυγή και την δαπάνη δημόσιου χρήματο, κανεί δεν διώχθη. Κανεί. Τίποτα το φοβερά αξιόπινο και κολάσιμο δεν ε, αποκαλύφθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει για το χρήμα που κρύβεται στην Ελβετία και σε άλλα μέρη του κόσμου και στη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό όχι γιατί υπάρχουν κάποιε φοβερά εγκληματικέ οργανώσει, αλλά είναι γιατί είναι ανίκανοι οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι φοβούνται την υπερφορολόγηση και να χάσουν την περιουσία του. Και η Deutsche Bank έχει πρόβλημα. Ε, ε, είναι και αυτό ένα καρφί στο ίδιο φέρετρο. Και ε, σκεφτείτε όλους αυτούς τους βοηθούς και συμβασιούχους του Ευρωκοινοβουλίου που δεν πληρώνουν φόρους. Φόρους δεν πληρώνουν και ευρωβουλευτές. Να η μεγαλύτερη φοροδιαφύγη του κόσμου. Πώς μου κάνετε όλοι εδώ τους ενάρετους ενώ είσαστε οι πρώτοι. Ε, η Ελβετία ίσως να γίνει κάτι σαν ε, ελληνική Βρετανία από τη δική μας πλευρά και να σας ε, βάλουμε εμείς ένα μαύρο κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Ποιοι είσαστε να αποφασίζετε ποιοι είναι οι φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρωπαϊκή ύπερο; ε, Είναι πολλοί αυτοί που έχουν κάνει και αυτοί οι δουλειές στις Ελβετίες και να πώς καταστρέφεται την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ε, δεν έχετε δικαίωμα να θέσετε φόρους σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η Βρετανία θα κάνει ό,τι θέλει μετά τον Brexit και ίσως να συνεργαστούμε με την Ελβετία και άλλες χώρες όπως τις κατεχόμενες Ουγγαρία και Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που απειλούνται και ε, πιέζονται διότι έχουν κάνει δηλώσεις και θέλουν να προασπιστούν την δική τους ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία να είστε ρεαλιστές. Οι Αμερικανοί δεν θα σας ανεχτούν, ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Απανατολοί. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσετε. Ποιο είναι το γαλλικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το γαλλικό μοντέλο ε, που είναι στραφοδιαβασμένο κιόλας. Διότι ούτε να ανταγωνιστείτε παγκοσμίως μπορείτε, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε οι τελευταίοι που θα φύγουμε. Είμαι βεβαίως ότι και οι Πολωνοί, και οι Τσέχοι και οι Ουγγροί ε, θα μα ακολουθήσουν. Και ίσω να δημιουργήσουμε έτσι μια διαφορετική ευρωπαϊκή διευθέτηση. Λίγο καλύτερη από αυτή που έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εμεί σα ευχαριστούμε. Και εγώ γερμανικά, αν μου επιτρέπετε. Πολύ σύντομα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές μας που ήρθαν από μακριά. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνατε διακινδυνεύοντας την ε, ε, υγεία σας και την καλή κατάσταση των παιδιών σας. Πολλά από αυτά που είπατε επιβεβαιώνονται και από τον ΩΣΑ. Αναφέρθηκαν ε, ε, γκρίζοι, μαύροι κατάλογοι και ε, πώς, ποιοι θα μπουν στους καταλόγους αυτούς. παίζει ρόλο το αν έχουν αρθεί τα πέντε επιζήμια καθεστώτα, όπως είπαμε. Ε, μετά από όλα αυτά, ε, μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη μετά από τη σημερινή συζήτηση ε, σχετικά με το τι θα γίνει, τι τύχη θα έχει η Ελβετία σε σχέση με τους καταλόγους. Εμείς, ε, ευχαριστώ για την ερώτηση, πρέπει να τηρήσουμε τη διαδικασία. Εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι για θέματα ε, επιζήμιο και αθέμη του φορολογικού ανταγωνισμού. Εδώ μιλάμε για καταγγέλλοντες, για μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε θέματα ξεπλήματος χρήματος. Αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα, τέλος του χρόνου, αρχές ε, του επόμενου έτους θα αποφασίσουμε αν θα μπει σε κάποιο κατάλογο η Ελβετία. Ε, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα συμμορφωθεί προς τα υπεσχημένα. Στη δέσμευση που ανέλαβε ε, αναφέρονται τα, μόνο τα πέντε επιζήμια καθεστώτα που πρέπει να καταργήσει. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ε, επίπεδο που είναι στο μέλλον. Εκεί θα εξετάσουμε αν η, τα νέα μέτρα για τους φόρους των επιχειρήσεων που ε, εισήχθησαν ως αντίμετρο αν αυτό Τέσσερι συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό θα γίνει σε ένα δεύτερο στάδιο. Και εκεί θα ληφθούν περισσότερα πράγματα υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε